Καλημέρα. Καθίστε παρακαλώ. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλωσορίζω και την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Καθίστε γιατί ακολουθεί μια μακρά ψηφοφορία. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο το καλύτερο. Καλωσορίζω την Επιτροπή Προπολογισμού και τον Πρόεδρο, τον κύριο Αχτιουή. Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω και τον συνεισηγητή, τον κύριο Ashworth. Θέλω απλώς να ανακοινώσω κάτι. Υπάρχει ένα ασφάλιμα στον κατάλογο ψηφοφορίας για το 183.2 είναι μια τροπολογία ΛΥΜΠΕ 17 στη σελίδα 20 περίπου του καταλόγου ψηφοφορίας υπάρχει ένα μείον στον κατάλογο, αλλά ο εισηγητής προτείνει συν αντί για μείον. Στο 183 σημείο 2, στην τροπολογία ΛΥΜΠΕ 17, ο κατάλογος ψηφοφορίας έχει μείον, αλλά ο εισηγητής προτείνει συν στη σελίδα 19 ή 20 αν θυμάμαι καλά. Η τροπολογία 17 της ΛΥΜΠΕ για το άρθρο 183 σημείο 2. Χάρη στους σκιώδεις συζητητές καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά για το θέμα. Μετά τη ψηφοφορία θα ξεκινήσει και η πραγματική δουλειά γιατί θα προσπαθήσουμε όλα αυτά τα οποία θα έχουν γίνει αποδεκτά να τα διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας. Ευχαριστώ τον κύριο Αχτουή, ο οποίος θα προεδρεύσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε και η Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές, τον Ρίτσαρντ Ασχουρθ και την ε, Ingeborg ε, Γκρέμπλε. Σας ευχαριστώ και τους κοιόδης ε, εισηγητές για μια τεράστια προσπάθεια που έκαναν για να καταρτιστούν οι κατάλογοι αυτοί των ψηφοφοριών χρειάστηκε να περάσουμε όλη τη νύχτα. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες από τη Γραμματεία που ήταν πάρα πολύ επιμελής. Είναι περίπλοκο το κείμενο. Πρέπει να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια απλούστευση. Ελπίζω να συνεισφέρουμε κι εμείς, όχι μόνο για τις, να συνεισφέρουμε στις υπηρεσίες της Κομισιόν και για το καλό των υπηρεσιών της Κομισιόν, αλλά και για τους ε, δικαιούχους. Έχουμε συνολικά 756 τροπολογίες. Κάποιες θα, τις, θα καταπέσουν, είτε γιατί δεν αφορούν την, ε, τις μικτές αρμοδιότητες των, τις αρμοδιότητες των ε, επιτροπών μας, είτε γιατί είναι αποκλειστική αρμοδιότητας άλλων επιτροπών που εμπλέκτηκαν ε, δυνάμει του άρθρου 54. Εάν δεν έχουν κάποιες δηλώσεις να κάνουν οι εισηγητές μας, τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Βάλτε σας παρακαλώ την κάρτα σας ε, στο ηλεκτρονικό κουτί για να κάνουμε μια διοκτημαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Καταγράφουμε 738 άτομα που ψήφισαν, 4 δεν έχουν ψηφίσει. Μόλις ήρθε και η κυρία Τωμά. 39 τώρα. Βλέπω μια στάθεια. Α, φτάσαμε στους 40. Ah, Νομίζω ότι εντάξει. Εντάξει τα νούμερα. Έχετε τους καταλόγους σας. κυρία Σολίν αλλάζει θέση. Ωραία, τα καταφέραμε. Τροπολογία 211, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 363, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 364 αποσύρεται. Η 365. Ψηφίζουμε τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Καταπίπτει. Πάμε στην 366 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 367 υπέρ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 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 27 ψήφοι 15 υπέρ. 3,91 υπέρ. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. 3,90 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 390. Ε, Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τη προφορίας. Απορρίπτεται. 27, 24 ψήφοι κατά, 18 υπέρ. 3.91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεβε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Είναι συμβιβασμό, έτσι. Θα το επαληθεύσουμε τώρα ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε 27 ψήφι υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 402 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 21 που θα μπορούσαν να ψηφιστούν μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετούνται. 403 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Άποχες υιοθετείται. 404 καταπίπτει. Και η 405. Πάμε στην 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα την επαληθεύσουμε. Την 22 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται 25 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Η 405 δεν καταπίπτει. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψηφίσουμε την 405. Ζητώ συγγνώμη που έκανα αυτό το λάθος και πάμε πίσω. Ποιος είναι υπέρ της 405. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. Δηλαδή. 406 και 407. 408, 409. Όλες μαζί υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι καταπίπτουν, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας Απορρίπτονται. 21 ψήφι υπέρ, 21 κατά. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 410 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 413 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 414 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 415 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 416 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 417 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 418 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 25. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορία Υιοθετείτε. 26 ψήφι υπέρ, 16 κατά. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 4-19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα την επαληθεύσουμε. Σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείται 25 ψήφι υπέρ, 18 κατά. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 420 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28 και 421 που είναι οι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.23 υπέρ. 4.24, 4.25 και 4.26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 427 και 428 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 30 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 429 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 430 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 431 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 433 υπέρ κατά αποχές θα τις επαληθεύσουμε χρονικά. Την 31 και 433. Πέρας φοφορίας. Υιοθετούνται 24 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. 4 4-34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι υπέρ, υπέρ, ε, υπέρση κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, άποχες. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα την επαληθεύσουμε. Θα την επαληθεύσουμε. 32 λοιπόν. Πέρας οφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία είχατε 33 υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται 4.35 υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι εγκρίνεται λίμπε 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.37 υπέρ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 Α, όχι, καταπίπτει. 4,41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4,42 υπέρ. Καταπίπτει, λάθος. 4,43. Επίσης καταπίπτει. 4,44 και 4,45 που έχουν τον ίδιο στόχο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 4,46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 447 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 448 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 449 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 450 και 452 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 451 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 453 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 454 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 455 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 4.56 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4.57 καταπίπτει. Πάμε στην 458 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 3α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 461 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 462 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίπε 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 και 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 465 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 464 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 466 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 467 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 468 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 469 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4,72 αποσύρεται. 4,73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαγγελθώσουμε ηλεκτρονικά. Τέσσερα ψηφίσουμε την 473 ηλεκτρονικά περισφοφορίας απορρίπτεται. 23 ψήφοι κατά με 20 ψήφους υπέρ. 470 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ομπλουά 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 474 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 475 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 476 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 477 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47, 478 είναι ίδιες, υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνουν όλα τα χέρια. Άρα ψηφίσουμε χρονικά τώρα. Πέρας φοφορίας. Υιοθετείτε. 27 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Αφέτ 8 υπέρ. Κατά θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 28 εναντί 14, 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αφέτ 9, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 479 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 480 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 481 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αγκρί 3 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίφθηκε. 482 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αγκρί 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 483 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 484 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Πεσ 4 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 54 υπέρ κατά Αποχές εγκρίθηκε. Πες πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 485 και ομπλούα 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 487 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 486 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά ε, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίφθηκε με 21 έναντι 17. Ρέτζι, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το ΙΡΕΤΖ 27, 488 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 56, 489 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 490 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Λίμπε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Λίμπε 13 υπέρ κατά εποχές εγκρίθηκε. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά Αποχέσα εγκρίθηκε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. 496 καταπίπτει 62 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίθηκε 63 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίθηκε 64 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίθηκε.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 εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73, τρία, ποιος είναι υπέρ, κατά. Δεν βλέπω πολλά χέρια που σηκώνονται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 και 77. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 505 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Από την 79 μέχρι την 89 έχουμε προτάσεις τροπολογιών ε, ε, διαγραφής που θα μπορούσαν ε, να ψηφιστούν μαζί, on block. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, περνάμε απευθείας στην 90, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 508 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 509 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 510 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 καλύφθηκε 92 511 μαζί ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 512 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 513 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 514 κατά πίπτη, 515 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 515. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 23 ψήφους έναντι 13, 516 κατά 517 ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 518 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 101 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 519 και 520 αποσύρθηκαν, 104, 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 521 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 522, 523 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 524 αποσύρθηκε, 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 525 αποσύρθηκε. ΔΕΒ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 και 526 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται 528 καταπίπτει εφόσον η 526 εγκρίθηκε. ΔΕΒ 7 και 527 υπέρ α, καταπίπτει 108 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 529 με, σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 530 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 531 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 532 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 533 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 534, 535, 536, 537, 538 και Ρέτζι 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Α, ε, καταπίπτει 539 καταπίπτει. Επίσης 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 ποιος είναι ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 540 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 541 καταπίπτει, 114 και 542 μαζί, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 543-544 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 14, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 545, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 547 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 548 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 551 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 552 αποσύρεται. 553 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 554 καταπίπτει. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 556 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 557 με ε, ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒ Εννέα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 558. Υπέρ, κατά, αποχές θα ε, παληθεύσουμε. 558 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 19 ψήφους έναντι 17. 560-559 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, Δευ 10. Όχι καλύφθηκε 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 561 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 562 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 563 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 564 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 505 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 566 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 568 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 569-570 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 571 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 572 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 573 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 575 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 574 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους εναντί 13, ΔΕΒ 12 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 130-576 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 577 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 578, 579 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 580 υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 21 ψήφους εναντί 15. 132. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 583. Ποιος είναι υπέρ, κατά, ε, ε απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 584 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. 585. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 ε, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 587 καταπίπτει, 588 αποσύρθηκε, 137, 589 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 17 με ευνοϊκή γνώμη των εισηγητών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αλλά θέλω να επαληθεύσω. πέρας της ψηφοφορία. εγκρίθηκε με 21 ψήφους έναντι 15. Συμβιβασμός, όχι, 590, 591, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, εγκρίνεται, 5, ε, εγκρίνεται, 139 ναι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 140 υπέρ, κατά, 141. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 595. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 598. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 13 υπέρ Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Βαίνει 599 πρώτα. Α, το ψηφίσαμε αυτό. Το ψηφίσαμε αυτό. Με συγχωρείτε. ΔΕΒ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 144 και 600 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 601, 602, 603 καλύφθηκαν

αποχές εγκρίνεται, 606 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 607 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 608 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 610 και 609 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 611 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δεύε 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6-12, 6-13 και Δεύε 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6-14, 6-15 και Δεύε 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6-16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6.17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6.18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 619, καλύπτεται. 6. Είναι συμβατή 619 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 620, 621 είναι οι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλει κάποιο το λόγο, θέλετε να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Την 620 και 621. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 ψήφοι υπέρ, 16, 21 ε, κατά 16 υπέρ. Ρέτζι 29. Όχι, όχι. Η Ρέτζι 29 συμπεριλαμβανόταν στις προηγούμενες. Η έμπλη 10 καλύπτεται 6-22 υπέρ. Κατά αποχές εγκλίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 623 υπέρ κατά καταπίπτει η 623 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 624 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 625 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 627-628 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 629 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 καταπίπτει, 630 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 631 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165-633 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 635 και Regi 31 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Ρέτζι 32. Όχι, η 636 και η έμπλη 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 32 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 17 κατά γιατί προσθέσαμε μία ψήφο, εγκρίνεται. Ρέτζι 32. 166 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 637 υπέρ... Α, όχι, καταπίπτει. 638 με μία προφορική τροπολογία υπέρ... Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 639 και έμπλη 12 υπέρ... Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 640 υπέρ... Κατά αποχές εγκρίνεται 6.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 642 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 643 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 644 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 648 υπέρ, κατά, Α, έχει αποσυρθεί, όχι δεν έχει αποσυρθεί, 648 Ζητώ συγγνώμη, 648 υπέρ, κατά, Έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. 171-172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 649 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 650, καταπίπτει. Συνδεστική λύση 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.56. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6.60. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΦΕΤ 16. Όχι, όχι. Συμβαστική, λύση, συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΑΦΕΤ 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΑΦΕΤ 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σηκώνετε το χέρι παρακαλώ με βολεύει 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 675 καταπίπτει 182 υπέρ Να ψηφίσουμε on block. Θα πρέπει να τις ψηφίσουμε χωριστά, συγγνώμη, 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές. 185 είναι ίδια, μπορώ να το... 186 ίδια, 187 ίδια, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Όλες αυτές εγκρίνονται. 676. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 203. 677 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 678 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 205 καταπίπτει, 22 καταπίπτει, 679 καταπίπτει, 206 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 207 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Αλλά παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας για να σας βλέπουμε. 207 υπέρ. Κάποιοι ακόμη δεν σηκώνουν τα χέρια τους. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 23 καταπίπτει. 681 καταπίπτει. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209 και λίμπε 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 682 καταπίπτει. 683 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 684 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 685 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 686 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 687 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 688 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 689 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 690 Έχουμε μία προφορική τροπολογία της κυρίας Χολμάγερ και μία τροπολογία του κυρίου Μάνκα που εγκρίνεται από την κυρία Χολμάγερ. Σωστά. Κυρία Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατόπιν συνεννοήσεως με την κυρία Χολμάγερ άλλαξε μια λέξη. Μιλάμε για τη διαδικασία έγκριση στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 258 Ήταν ένα λάθος το οποίο διορθώθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 694 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, στη συνέχεια έχουμε κάποιες ε, όπου μπορούμε να έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα. Ας περάσουμε λοιπόν στη σελίδα 75. Διορθώνω στο κάτω μέρο τη σελίδα 74, τροπολογία 754. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 754 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 755 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 756 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αφέτ 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. 213 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έσ, 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 215 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 216 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 217 και αφέτ 1 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. 2.18 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Δεύε 1 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2.19 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2.20 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2.21 υπέρ, κατά, αποχές να το επαληθεύσουμε την 221 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται σαφώς 26 ψήφοι κατά. Αν σηκώνετε το χέρι θα είχαμε αποφύγει την ηλεκτρονική 2.22 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 2.23-2.24 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2.25 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2.26 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Αφέτ 2 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2.28 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2.27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αφέτ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 2 με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 2 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε για τη Ρέτζι 2 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 ψήφοι κατά 16 υπέρ 2.39 υπέρ κατά δεν βλέπω να σηκώνει κανείς το χέρι αποχές απορρίπτεται 1 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αφέ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.43 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται ή όχι. Έχετε δίκιο, εγκρίνεται. 2.53, 2.54, 2.55 και 4 της Reggie 4 ήταν κομμάτι της ίδιας και εγκρίνεται. 2.56 με αρνητική ε, πρόταση ε, του εισηγητού υπέρ, κατά, να επαληθεύσουμε. 2.56. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 23 κατά. 2.59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αφέτ 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές να επαληθεύσουμε τη 283 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Ρέτζι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 286 υπέρ. Με μια προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 289 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 10 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 22 ψήφοι κατά 15 υπέρ. 2,92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.93 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.95 απο, ε, αποσύρεται. 2.97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 11 και 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 2.98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 301-302 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 304-305 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 306 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 307-308 υπέρ, κατά αποχές 300, απορρίπτεται 310-311 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 312-313 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 314-315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 323 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, υιοθετείται, διορθώνει Πρόεδρος. 327, 328, 329, 330. Και η τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται. Πες 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 334-335 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ρέτζι 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζο 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 336 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζο 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζο 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 22. Τελικά θα ψηφίσουμε τη Ρέτζι 22. Να, από ό,τι φαίνεται. Ψηφίσουμε τη Ρέτζι 22 υπέρ. Κατά. Μου είπαν ότι είναι λάθος. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, άρα πρέπει να την ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία της Ρέτζι 22. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Όμπλου 3 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 339 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 345 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 346 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Πολύ ωραία. Πάμε στην ψήφιση της έκθεσης όπως την τροποποιήσαμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ, μία αποχή όχι, 13 εποχέ, λέει ο πρόεδρο. Θερμά συγχαρητήρια στους ηγητές. Και τώρα πρέπει να πάρουμε θέση για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε μια ονομαστική κλίση. Ξεκινάει η σφοφορία τώρα. Χρειαζόμαστε μια πλειοψηφία 36 ατόμων, 36 ψήφων για την εντολή. Αλλιώς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τώρα ψηφίζουμε για την εντολή. Διάφορες συζητήσει εκτό μικροφώνου. Τι ψηφίζουμε ακριβώς. Ψηφίζουμε για πρόεδρο την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε τώρα. Κάποιοι δεν ψήφισαν ακόμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Έγκριση με 30 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και 13 εποχές. Ωραία. Και τώρα θα πρέπει να πάρουμε θέση επί της εντολής για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Πρόκειται για την εφαρμογή του, κανο... του άρθρου 69C που απαιτεί μία πλειοψηφία των βουλευτών της Επιτροπής μας, της Μικτής Επιτροπής. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε 36 ψήφους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Είμαστε 70 όλοι όλοι, 40 η κοντ, οι άλλοι 30. 35 είναι, είναι οι μισές ψήφοι, η πλειοψηφία είναι 36 ψήφοι επομένω. Είναι για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, έτσι. Δεν αποφαινόμαστε, δεν υιοθετούμε ή όχι την πρόταση της Κομισιόν όπως την τροποποίησαμε. Ψηφίζουμε τώρα για την εντολή. Πέρας φοφορίας. 43 ψήφοι υπέρ. Δίδεται η εντολή. Είχαμε προβλέψει ότι θα τελειώσουμε αυτή τη ψηφοφορία πριν τις 11. Το καταφέραμε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Σας παρακαλώ, ακούστε μας. Δεν τελειώνει εδώ η συνεδρίαση. Η κυρία Γκρέσλα έχει την, το λόγο. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού τώρα θα συνεδριάσει στην 5G3. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα, ξεκινήσει τη συνεδριασή της στις 11 η ώρα σε αυτή την αίθουσα η κοινή συνεδρίαση